Chers collègues, bonjour. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σε αυτή την τελευταία ημέρα της Ολομέλειας που ως συνήθως τις Πέμπτες στο Στρασβούργο συμπίπτουν πολλές συνεδριάσεις. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Τρομοκρατία και θα σα πρότεινα να περάσουμε αμέσως στο σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης και να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, να, τις, να την εγκρίνουμε. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων της 5ης, 11ης και 12ης Ιουλίου 2018. Αν δεν υπάρχουν και εδώ αντιρρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά. Σημείο 3 ανακοινώσεις. Ως συνήθως. Καταρχήν θα ήθελα εν είδη εισαγωγής να σας ενημερώσω ότι η συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου αναβα... ακυρώνεται. Κανονικά θα έπρεπε να αφιερωθεί στην εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών με τα από την προεργασία που έκαναν ε, οι συνεισηγήτριες και οι σκιώδεις αλλά επειδή κολλείεται μια συνεισηγήτρια για τις 15 Οκτωβρίου, προτιμήσαμε να ακυρώσουμε τη συνεδρίαση, αναζητώντας μια άλλη πιο βολική ημερομηνία. Επίσης, να σας ενημερώσω στις ανακοινώσεις ακόμη, ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής ΤΕΡ συμμετείχαμε την άδεια της διάσκεψης των πρόεδρων και τηρώντα τη διαδικασία στην αποστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών στη Washington 16 με 19 Ιουλίου με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορούσε και τη δική μας Επιτροπή. Συμμετείχα σε πολύ σημαντικές συναντήσεις ε, με θέμα τη συνεργασία με τους εταίρους μας ε, πέκνα του Ατλαντικού στον τομέα της τρομοκρατίας και εκπονώ και μια σύντομη έκθεση για τα βασικά στοιχεία αυτών των συναντήσεων που θα σας ενδιαφέρει και θα σας μοιραστεί όσο νούπο. Αυτά ως προς τις ανακοινώσεις και περνάμε στο κυρίως θέμα της σημερινής μας έκτακτης συνεδρίας, γι' αυτό άλλωστε και έγινε είναι το σημείο 4 που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με τον Sir Julian King, που είναι ο αρμόδιος επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητέ Sir Julian, νιώθουμε μεγάλη χαρά και τιμή που έχουμε την ευκαιρία να σας ε, ξαναφιλοξενούμε στην Επιτροπή μας γιατί το χαρτοφυλάκιό σας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μαζί με τον Επίτροπο είχαμε ήδη εγκαινιάσει τις εργασίες της Επιτροπής μας τον περασμένο Οκτώβριο και ήδη από την ε, αρχή, από τη σύσταση της Επιτροπής μας, είχαμε την αμέριστη υποστήριξη και με και συνεχή διάλογο με τον ε, Επίτροπο Κίνγκ. Και όλους αυτούς τους μήνες ε, συνεργαστήκαμε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και μάλιστα ήταν ε, ε, σημαντικό και δεικτικό και συμβολικό να ξανακαλέσουμε τον Επίτροπο σε αυτή την σχετικά προχωρημένη φάση και λίγο πριν την διεκπαιρέωση των εργασιών μας να ξανακαλέσουμε τον Επίτροπο για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο με σας κύριε Επίτροπε προγραμματίζοντας αυτή την ανταλλαγή απόψεων γιατί είστε ο στενότερος ε, και από τους πιο αξιόπιστους εταίρους μας και συνεργάτες ε, σε αυτή τη προσπάθεια. Ε, και το λέω έτσι για να μην κακοκαρδίσω κανέναν άλλον συνεργάτη και εταίρο. Είμαστε ευγνώμων, το καταλάβατε και από τα χειροκροτήματα. Δεν, δεν πρόλαβε καν να μιλήσει ο Επίτροπος. Ίσως μετά δεν έχουμε τέτοιες επιφημίες. Πάντως ενδιαφέρον θα ήταν, αν συμφωνείτε και εσείς με την αρχή κύριε Επίτροπε, πρώτα να μας κάνετε μια σύντομη ενημέρωση για τα βασικά θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μας κατατοπίσετε για τα μέτρα που εξετάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα σε ζητήματα αντιτρομοκρατίας και επίσης μια και από τους ε, πρώτους παραλήπτες του σχεδίου έκθεσης της Επιτροπής μας να μας πείτε και τη δική σας γνώμη αν έχετε παρατηρήσει ή σχόλια επί του σχεδίου έκθεσης. Όπως ξέρετε, προκάλεσε την ιδιαίτερη προσοχή και το ζωηρό ενδιαφέρον ε, όλων των συναδέλφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μάλιστα έχουν κατατεθεί αυτό το σχέδιο έκθεση 1520 τροπολογίες. Οπότε, στα πλαίσια αυτής της εξαιρετική συνεργασία που έχουμε, καλό θα ήταν να μας παρουσιάσετε και τη δική σας θέση και απόψεις για αυτό το προκατακτικό σχέδιο έκθεσης. Και πριν σα δώσω το λόγο, κύριε Επιτροπέ, θα διαπιστώσατε στην έκθεσή μας ότι ομόφωνα προτείνουμε να διατηρηθεί αυτό το ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή το χαρτοφυλάκιο της Ένωσης Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη νέα θητεία της. Δεν θα μακρηγορήσω λοιπόν, αγαπητέ Επίτροπε. Σας δίνω τώρα και κάποια εισαγωγικά σχόλια και θα σας πρότεινα να μην ξεπεράσετε το τέταρτο στην αρχική σας αυτή ομιλία και μια και έχετε εξοικειωθεί με αυτή τη διαδικασία, μετά την δική σας ομιλία θα έχουμε τη διαδικασία ping-pong ερώτα με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Members, και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ πολύ. Ε, ξέρω ότι θα σας απογοητεύσω πίνω καφέ και όχι τσάι. Αλλά πολύ ευχαρίστως και στο πνεύμα της χώρας που γνωρίζω καλύτερα ε, προσωπικά να παίξουμε και το πινκ pong όπως προβλέπετε στη συζήτηση. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την πρόσκληση, για την γενική υποδοχή στην Επιτροπή σας και για τη σημερινή συνεδρίαση που ξέρω ότι σας πιέζει γιατί υπάρχουν παράλληλα και άλλες ε, συναντήσεις ε, και υποθέσεις. Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Πριν από 12 μήνες μόλις με, με είχατε προσκαλέσει μια πρώτη συνεδρίαση. Πολλά όμως έχουν το μεταξύ συμβεί. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω μερικά λόγια για το παρελθόν αλλά και τα νέα ζητήματα που έχουμε στον τομέα της ασφάλειας ε, προωθήσει. Ξεκινώντας όμως θα ήθελα να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου για τη δική σας τη δουλειά των τελευταίων μηνών την οποία θεωρώ ευπρόσδεκτη, διάβασα το σχέδιο της έκθεσης. Ομολογώ βέβαια ότι δεν έχω διαβάσει κάθε μία τροπολογία χωριστά, αλλά ε, μια αρκετά μακροσκελή σύνοψη των τροπολογιών τη διάβασα και νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι έχετε την ε, ε, μεγάλη προσήλωση και ότι καταγράφεται μεγάλη προσήλωση και στράτευση στα θέματα αυτά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, στο επίπεδο της Επιτροπής σας βλέπω δηλαδή ότι με πολύ μεγάλη πρόσοχη επεξεργάζεστε τα θέματα αυτά. Και θα επανέλθω μετά. Το τελευταίο λοιπόν το δεκάμινο ακολουθήσαμε μία διτή προσέγγιση για να βελτιώσουμε τα ζητήματα ασφάλειας από τις απειλές, κυρίως τις προερχόμενες από την τρομοκρατία, δηλαδή τους τομείς τους οποίους ε, μπορεί να δράσει ο τρομοκράτης, ο οποιοδήποτε άλλος θέλει να κάνει κακό. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την αντοχή των συστημάτων και την προληπτική δράση και σε μία πρώτη προσέγγιση προσπαθούμε να περιορίσουμε την πρόσβαση των τρομοκρατών είτε σε ελεύθερη διακίνηση, είτε σε κυκλοφορία νομίσματος, είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε σε ε, εξοπλισμούς να περιορίσουμε την ελεύθερη διακίνηση ε, στα σύνορα, την χρήση πολλαπλών ταυτοτήτων με καλύτερη συνεργασία των συστημάτων ε, πληροφοριών, να ενισχύσουμε την ασφάλεια των εξωτερικών μας σύνορων όπου χρειάζεται ιδιαίτερα να καταπολεμηθούν προσπάθειες ε, αξιοποίησης της μετανάστευσης και της περί τη μετανάστευση τον περί μετανάστευση ζητημάτων και αξιοποίησης τους βέβαια για λόγους τρομοκρατικούς ή σύγχυσή τους. Ε, επίσης, τα δεδομένα, οι πληροφορίες έχουν κέρια σημασία για όλη αυτή την προσπάθεια. Ε, επιχειρούμε λοιπόν τη μεγιστοποίηση των ε, πλεονεκτημάτων που μας προσφέρουν τα συστήματα πληροφοριών εξασφαλίζοντας μια διαλειτουργικότητα που είναι το καλύτερο δυνατό και βέβαια καλύπτοντας ό,τι κενά μπορεί να υπάρχουν, συμφωνώντας ενδεχομένως σε νέα συστήματα πληροφοριών όπως το ETIAS, ε, το iCris ε, να ενδυναμωθεί και άλλα. Ταυτόχρονα ενισχύοντας και το σύστημα πληροφοριών Schengen και την ε, EU LISA που έχει τεράστια σημασία. Στο οικονομικό να είναι πιο δύσκολη δηλαδή η διάθεση χρημάτων από τους, ε, ε, από τους τρομοκράτες. Η πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομοποίησης παρανομών εσόδων έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί παρεμποδίζει την ε, χρήση αυτών των κονδυλίων. Η δική σας έκθεση έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την ανείχνευση προτάσεις. Ξέρω συζητήσατε και με τις Ηνωμένε Πολιτείες τα θέματα αυτά. Επίσης ένα συμπληρωματικό σύστημα ευρωπαϊκό υπό εξέταση αυτή τη στιγμή, το οποίο και προσωπικώς εγώ ε, υποστηρίζω, γιατί θεωρώ ότι προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ε, στα θέματα των όπλων έχουμε τις προτάσεις για τον περιορισμό εισαγωγών-εξαγωγών, ώστε να μην υπάρχει διαθεσιμότητα του υλικού εκείνου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ε, είτε είναι πυρομαχικά είτε είναι όπλα για την κατασκευή επί παραδείγματι βομβών. Περιορισμός της πρόσβασης σε ανθρώπινο δυναμικό, αυτούς προσπαθούν να επιστρατεύουν, προσπαθούμε δηλαδή να περιορίσουμε την ριζοσπαστικοποίηση είτε μέσα στις κοινότητες, σε όρους ε, συμμετοχής σε μια κοινότητα, είτε διαγραμμικά, γιατί η διαγραμμική πρόσβαση και ε, πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ε, τρομοκρατικές επιθέσεις όπως έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Και βεβαίως περιμένω και τις δικές σας τις προτάσεις. Στο σχέδιο έκθεσης επίσης δίνεται μεγάλη προσοχή στο θέμα των θυμάτων, πολύ σωστά, πώς θα τα βοηθήσουμε. Συμφωνώ απολύτως και σε αυτό. Από πλευράς της Επιτροπής ε, για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της τρομοκρατίας και Καταρχά, σε πρώτο στάδιο και βέβαια τα υπόλοιπα μπορούμε να τα δούμε και στο, στη φάση των ερωτήσεων και αποκρίσεων, αλλά σε πρώτη φάση πρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό το οποίο έχουν συμφωνήσει να πράξουν. εφαρμόζοντας δηλαδή τα μέτρα που προβλέπει η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας γιατί πολύ λίγα είναι τα κράτη-μέλη τα οποία μέχρι τώρα έχουν ε, εισαγάγει στην εθνική νομοθεσία αυτή την οδηγία, που αποτελεί και εκτιμένο. Επίσης, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος, η προστασία των δημοσίων χώρων πρέπει να βελτιωθεί, οι παράγοντες που έχουν δημόσια δράση, είτε είναι ιδιωτική είτε είναι ε, δημόσιο, πρέπει να συνεργαστούν, ε, εναέριες στις μεταφορές περιορισμός των κινδύνων από πυρηνικές, βιολογικές, χημικές, ε, μικροβιολογικές ε, απειλές, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε κι εσείς, κίνδυνος αφηρημένος μεν πολύ ε, πραγματικός δε εάν επί δούμε το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, κύβερνο επιθέσεις Εδώ και είναι συγγραφέ με όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα. Ο κ. Γιουνκέρ και στην ομιλία του για την κατάσταση ένωση ε, την περσινή είχε πει ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα για την καταπολέμηση των κυβερνών απειλών. Έκτοτε, μέσα αυτό το δεκάμινο δηλαδή, και σε συνεργασία πιστεύω μαζί σα, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο για μια νέα στρατηγική κυβερνό ε, που στηρίζεται και στην ενίσχυση της ε, ανθεκτικότητας των αμυνών, τη συνεργασία για την κυβερνοάμυνα και βλέπω ότι όλο το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την ε, πρόθεση για την θέσπιση μιας νέας υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας. Προτάσεις επίσης για μέτρα αντιμετώπισης είτε απόκρυψης, της απόκρυψης πληροφοριών είτε των ψευδών πληροφοριών, των fake news, ε, ή ό,τι άλλο μπορεί να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο επίση πρέπει να αναλυφθούν. Επίση, ο πρόεδρος Γιούνκερ φέτο μίλησε για νέε εξελίξει στη δουλειά που θα κάνουμε από κοινού. Αφενός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση για καλύτερη αντιμετώπιση του τρομοκρατικού περιεχομένου που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο όπω ανέφερα μόλι τώρα κάθε μία από τις επιθέσεις, δηλαδή την οποία έχουμε μέσα το τελευταίο 18 μήνο ή τη διετία αντιμετωπίσει, είχε και διαγραμμικό στοιχείο. Μέσα από το διαδίκτυο, παραδείγματι, κυκλοφορούσαν είτε προαγωγή της ιδέας της τρομοκρατικής ή ακόμα και οδηγίες για μια τρομοκρατική επίθεση ή γενικά ε, καθοδήγηση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ένα φαύλο κύκλο, ε, τον οποίο πρέπει να σπάσουμε, γιατί, πλήτη, γιατί απευθύνεται βέβαια σε νεότερου συνήθω ανθρώπου. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το πόσο το υλικό αυτό της ε, καθοδήγηση τρομοκρατικής των οδηγιών μένει πάνω στο διαδίκτυο. Τα τρία τέταρτα των συνδέσμων, για παραδείγματι, της ε, προπαγάνδας της, ε, της ίσης, μέσα σε τέσσερι ώρες έχουν κυκλοφορήσει, έχουν μοιραστεί από τον ένα στον άλλον. Γι' αυτό η ταχύτητα έχει τεράστια σημασία στην αντιμετώπιση αυτών των απειλών και γι' αυτό προτείνουμε νέα νομοθετήματα στον τομέα αυτό. Έχουμε σε οθελοντική βάση παρακολουθήσει μία πρόοδο στις πλατφόρμες η οποία είναι αρκετά ικανοποιητική αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και προτείνουμε πρώτον να είναι υποχρεωτικό κάθε πλατφόρμα να αντιδρά μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που θα λάβει εντολή διαγραφής ε, περιεχομένου από δικαστικές ή αστυνομικές αρχές όταν πρόκειται για καθαρά τρομοκρατικό περιεχόμενο. Δεύτερον, Εάν μια πλατφόρμα αποδεδειγμένα αξιοποιείται από τρομοκρατική οργάνωση για τη διάδοση αυτού του περιεχομένου, οι αρχές του κράτους μέλους και η εν λόγω πλατφόρμα θα είναι, θα είναι υποχρεωτικό να κάτσουν και να συζητήσουν μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης ε, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται το περιεχόμενο, να μην επανεμφανίζεται με σαφείς κανόνες και ε, διασφαλιστικές δικλείδες ή καλύτερα σαφέστερους κανόνες και διασφαλιστικές δικλείδες από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και τρίτον και πολύ πιο σημαντικό, θέλουμε τα κράτη-μέλη να ε, έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν, να προβλέψουν επαρκείς ε, επαρκές δυναμικό και ικανότητες ε, εφαρμογής και επιβολής του νόμου, αστυνομικές δηλαδή δυνάμεις, για την καταπολέμηση αυτού του κινδύνου της ε, διάδοσης τρομοκρατικού υλικού στον κυβερνοχώρο. Κάποια κράτη το έχουν κάνει, όχι όλα, χρειαζόμαστε περισσότερες προσπάθειε. Επίση, άλλε διασφαλιστικέ δικλείδε, αποτελεσματικό μηχανισμό για την κατάθεση προσφυγών ή επισήμανσης προβλημάτων και αστυνομική συνεργασία βεβαίως. Όλα αυτά σημαίνουν ότι κάπου μπορούν να υπάρχουν κάποιες δυνατότητες που άλλοι ίσως να μην ε, προβλέπουν και γι' αυτό θέλουμε να συμφωνήσουμε τα κράτη-μέλη κατόπιν προτάσεών μας ε, για την επιβολή κυρώσεων εάν κάποιο δεν συνεργάζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν αντιδράσει αμέσω σε μια περίπτωση θα επιβάλλονται ε, κυρώσει. Αλλά εάν, παραδείγματι, μια πλατφόρμα συστηματικά δεν συμμορφώνεται, τότε θα προβλέπονται ουσιαστικέ κυρώσεις οι οποίε μπορεί και να φτάνουν μέχρι τον, ε, το κλείσιμο με βάση και τους κανόνες που έχει ο κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, οι εκλογικέ διαδικασίες που μας περιμένουν. Οκτώ συνολικά στην προσεχή περίοδο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και βέβαια και οι ευρωεκλογέ. Έχουν τη συνάφειά τους εδώ χωρίς εγώ να έχω στη μου στοιχεία συγκεκριμένα που να δείχνουν ότι μπορεί κάποιος να προβλέπει, να σκοπεύει, να πλήξει ή να επηρεάσει η εκλογική διαδικασία, αλλά με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα νομίζω ότι οφείλουμε προληπτικά να προετοιμαστούμε για μια τέτοια πιθανότητα. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις. Πρέπει να θεσπίσουμε τα μέτρα εκείνα τα οποία θα μας επιτρέψουν να είμαστε πιο ανθεκτικοί σε επιθέσεις τέτοιου χαρακτήρα ώστε να καταστεί πιο δύσκολο για τον οποιονδήποτε ενδεχομένω να ήθελε να ε, παρεμβεί ή να επηρεάσει ή να νοθεύσει αυτό το αποτέλεσμα. Επομένω, έχουμε την πρόθεση για καλύτερη συνεργασία, να πιέσουμε τα κράτη-μέλη για ένα εθνικό σύστημα συνεργασία εκλογική, αρμόδιε αρχέ, ε, φορευτικέ επιτροπέ, αρχέ κυβερνοάμυνα, ε, Επιβολή του νόμου αστυνομικέ αρχές κτλ. και συνεργασία σε ένα ε, ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο προετοιμασία των εκλογικών αναμετρήσεων και προστασίας τους. Επίσης με διαγραμμική ε, διαφήμιση ε, μπορούμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη τα συστήματά τους να προστατευθούν περισσότερο μπορούμε με τη διαγραμμική διαφήμιση να προειδοποιήσουμε τον κόσμο, 15-16 ε, Οκτωβρίου, όπως ξέρετε, έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση και είστε και ευπρόσδεκτοι. Εκεί θα συμμετάσχουν ε, διάφοροι φορείς ε, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα από όλα τα κρατημέλη. Οι δύο αυτές προτάσεις λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να λάβουν προτεραιότητα για να οδηγηθούμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα στο επόμενο δίμηνο, δεδομένου ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη θέσή μας. Πρέπει να εγκριθούν δηλαδή πριν να λήξει η τρέχουσα θητεία και βουλευτική περίοδος ε, και θέλουμε όλα αυτά να κλείσουν πριν το τέλος της θητείας. Και θέλουμε αποτελέσματα και στην άλλη νομοθετική πρόταση που έχουμε από κοινού επεξεργαστεί το τελευταίο, τους τελευταίους μήνες. Μια πολύ σημαντική πρόταση όπου εάν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τις διάφορες προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα ιδιαιτέρω σε κάθε πρόταση βεβαίω, αλλά η διαλειτουργικότητα που μα απασχολεί έχει τεράστια σημασία. Αυτό μπορεί να αφήσει ανοιχτό πεδίο ώστε να μα πλήξουν όσοι είναι κακόβουλοι. Ιδιαίτερη έμφαση νομίζω δίνει και η δική σας η έκθεση, το σχέδιο εκθέσεως, στην εφαρμογή της ήδη εγκριθής σας νομοθεσίας και βέβαια πρέπει να εξασφαλιστεί πρόοδο και στι προτάσει που είναι υποσυζήτηση. Ιδιαίτερα εσεί επιμένετε στην υλοποίηση όμω τη ήδη εγκριθής σα νομοθεσία. Άλλη μια μεγάλη πρόκληση που πρέπει από κοινού και με τα κράτη-μέλη βέβαια να αντιμετωπίσουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις ε, σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδο, αλλά σε άλλε. Δυστυχώ βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμη μεγάλο περιθώριο βελτίωση και πρόοδου και αυτό δεν πρέπει να το ε, λησμονούμε και να το παραγνωρίζουμε. Ε, το κομμάτι που έχει να κάνει με την οδηγία για τα μητρώα ονομάτων έχει πολύ μεγάλη σημασία. 17 κράτη-μέλη ήδη έχουν προχωρήσει σε πλήρη εφαρμογή, ακόμα δύο προχωρούν, αλλά πολλά είναι τα κράτη-μέλη που πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους σε αυτό. Επίσης, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πλήρη υλοποίηση μέτρων όπως η οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και ε, συστημάτων πληροφοριών οδηγία νης, όπου Λίγα μόνο είναι τα κράτη-μέλη που έχουν κοινοποιήσει εφαρμογή. Για την αστυνομία επίσης η άλλη οδηγία που μόνο ένα τρίτο των κρατών μέλων έχει κοινοποιήσει ε, εφαρμογή ή ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο. Άρα σε πολλά πεδία έχουμε να βελτιωθούμε. Και επίσης υπάρχουν και άλλα μέτρα των οποίων μόλις έληξαν οι προθεσμίες, καταρχάς ε, κατά πολέμηση τρομοκρατίας που ήδη ανέφερα και με την ε, εκπνοή της προθεσμίας τον προηγούμενο μήνα σημειώθηκε ότι μόνο πέντε κράτη-μέλη είχαν κοινοποιήσει πλήρη ενσωμάτωση και εφαρμογή. Αυτό για μένα είναι μια μεγάλη πρόκληση ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα. Όλοι ξέρουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η οδηγία. Πρέπει όλα τα κρατημένα λοιπόν να προχωρήσουν σε εφαρμογή. Και το άλλο θέμα που ξέρω ότι σας έχει επίσης απασχολήσει, σημαντικό αν και αμφιλεγόμενο σε ορισμένες χώρες, η οδηγία περί πυροβόλων όπλων. Τρία μόνο μέλη, έχουν κοινοποιήσει πλήρη εφαρμογή της οδηγίας αυτής, δεν αρκεί προφανώς, γιατί όλοι έχουμε συμφωνήσει ανεξάρτητος του θέματος στο οποίο κινούνται οι συζητήσεις ότι πρέπει να προχωρήσει η υλοποίηση αυτής της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα. Συνεχίζουμε λοιπόν, όλοι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ξέρω ότι με τη λήξη της θητείας έχετε πολλά ζητήματα να κλείσετε, πολλά έχετε να κάνετε κι εσείς από πλευρά σας. Ε, λίγος ο χρόνος που μένει Ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο εγώ έχω συνείδηση της χρονικής πίεσης ε, που έχω και εγώ να αντιμετωπίσω. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου πάντως ε, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να κλείσω τα θέματα και μαζί με εσά να ορίσω ένα πλαίσιο χρονικό για το επόμενο διάστημα. Που πιστεύω ότι θα είναι και το κύριο πλεονέκτημα της έκθεσης και της δουλειάς που κάνετε, δηλαδή ο προσδιορισμός ενός πλαισίου χρονικού που θα ορίσει τα επόμενα βήματα για το προσεχέ κοινοβούλιο, για την προσεχή ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν μου επιτρέπετε ένα προσωπικό σχόλιο, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η προσεχής Επιτροπή, ανεξαρτήτως της σύνθεσής της, να προβλέψει επαρκείς πόρους για τα θέματα της ασφάλειας. Νομίζω ότι μπορώ να το πω αυτό ελεύθερα γιατί δεν θα με αφορά προσωπικά. Αλλά οπωσδήποτε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά και πολλού τομεί στου οποίου θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε αποτελεσματικά από κοινού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε, για αυτή τη ε, συνθετική παρουσίαση, τις προοπτικές που μας δώσατε, για την ανάλυση που κάνατε, χωρίς να κάνετε καμία παραχώρηση σε σχέση με αυτά που έχουν αναγγελθεί, σε σχέση με αυτά που καμιά φορά καθυστερούν να εφαρμοστούν Σα ευχαριστώ για τι προοπτικέ και τι προτεραιότητες που αναφέρατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρουμε και τον ρεαλισμό σας και τον πραγματισμό σας, που τα διαπιστώσαμε και σήμερα το πρωί. Να δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα απ' όλα στην Helga Stevens, την συνεισηγήτριά μας, που ε, θα σχολιάσει. Ενδεχομένω να σας κάνει και ερωτήσεις. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την αναλυτική παρουσίασή σας, πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρον ε, τα πεπραγμένα σας και την ε, σαφή παρουσίαση των πεπραγμένων των κρατών μελών για τις διάφορες ε, οδηγίες, δηλαδή την εφαρμογή τους την μεταφορά τους και φαίνεται ότι ακόμη καθυστερεί και αυτό είναι λυπηρό. Όπως μας είπατε, τόσα κράτη-μέλη κολλησιεργούν. Δεν εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφόσον πρόκειται για θέματα ασφάλειας, μου είναι εντελώς αδιανόητο. Γιατί υπάρχουν τόσα κράτη-μέλη που στην ουσία ε, θέτουν εν κινδύνο την ζωή των ε, πολιτών τους. Γιατί το κάνουν, έχετε κάποιο λόγο, ε, είναι οικονομικό θέμα, είναι ότι υπάρχουν πολλές οδηγίες που πρέπει να μεταφερθούν και καθυστερεί η εφαρμογή τους. Ίσως χρειάζονταν κάποια κράτη-μέλη περισσότερη βοήθεια, ενδεχομένως και οικονομική, για να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία ή έχουν ε, άλλο χαρακτήρα οι λόγοι. Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι που τόσα κράτη-μέλη ακόμη δεν εφαρμόζουν αυτές τι οδηγίες, γιατί δεν συνεργάζονται ενδεχομένω ε, για θέματα ασφάλειας. Γιατί όλοι θα ωφελούνται από μια συνεργασία. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί τόσα κράτη-μέλη δεν συνεργάζονται. Για τον Οργανισμό Καταπολέμησης των Απατών ακούμε ότι θα αυξηθούν οι αρμοδιότητές τους. Και ορισμένοι λένε ότι θα έπρεπε να εμπλακούν και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αν υπάρξουν ε, προτάσεις ε, επέκτασης ε, της αρμοδιότητας του οργανισμού αυτού, φοβάμαι ότι δεν θα περάσουν από το Συμβούλιο. Γιατί λοιπόν να μπούμε στον κόπο να το επιχειρήσουμε. Έχω κάποιες αμφιβολίες και για την ενδεχόμενη προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας προσπάθειας. Οι εθνικοί πυρογνώμονε και οι εισαγγελείς ε, δεν μοιάζει πραγματικά να το επιδιώκουν και να, το, και να επιθυμούν να γίνει. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε τους ε, προηγούμενους μήνες, ελπίζω να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες και σας ευχαριστώ πολύ και για την δική σας προσωπική συμβολή στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Α, ναι, πινκ πονγκ, βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ για την εργασία σας ε, ως ε, Τώρα, η εφαρμογή. Συμφωνώ, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα. Νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες, και σε αυτό συνέβαλε και η έκθεσή σας, επιτύχαμε να έχουμε τις ε, μηνιαίες ε, εκθέσεις για την ασφάλεια στην Ένωση, αλλά και η συνεδρίαση η δική σας ε, τονίζει ότι υπάρχει καθυστέρηση. Στην τελευταία έκθεση για την ασφάλεια στην Ένωση που θα δημοσιευθεί στην, την επόμενη εβδομάδα, εξετάζουμε οδηγία, που υπάρχουν κενά στην εφαρμογή της κάθε οδηγίας, που έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες επί Πού πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Και κατά τις επισκέψεις μου στα διάφορα κράτη-μέλη, συστηματικά θέτω αυτά τα θέματα, όπου έχω πρόβλημα με την εφαρμογή από κάποιο κράτος μέλος. Και σας ενθαρρύνω και εσάς να κάνετε κάτι τέτοιο. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί περισσότερη δημοσιότητα στα κενά αυτά. Γιατί προκύπτουν τώρα. δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμη κακή θέληση. Αλλά κάποια κράτη-μέλη έχουν περισσότερες δυσχέρειες από άλλα για να εφαρμόσουν όσα έχουν αποφασιστεί. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να γνωστοποιούμε κάποια θέματα, να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να σημειώσουν πρώτα, αλλά πρέπει και να βοηθήσουμε και το κάνουμε με διάφορους τρόπους. Ως Επιτροπή τους δίνουμε τεχνικές συμβουλές, σε κάποιες περιπτώσεις και χρηματοδότηση. Άρα προσπαθούμε να διευκολύνουμε και τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ ομοτήμων δηλαδή. Γιατί κάποια κράτη-μέλη ε, αναπόφευκτα έχουν προχωρήσει περισσότερο από άλλα. Θα θέλαμε λοιπόν ε, πρωτοπόροι να βοηθήσουν τους βραδιπορούντες με διάφορα μέτρα και μέσω της πολιτικής στήριξης που και εσείς μπορείτε να τους δώσετε για να υπάρξει περισσότερη συνειδητοποίηση, ευαισθητοποίηση και ελπίζω μέχρι το τέλος ε, της θητείας μας να είναι πολύ καλύτερη η εφαρμογή για αυτές τις τόσο βασικές οδηγίες. για τον επόπτη προστασίας δεδομένων. Όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούγκερ στην ε, περσινή του ομιλία την κατάσταση της Ένωσης και κοιτάζοντας προς το μέλλον, σωστό λοιπόν που το αντιμετωπίζετε εσείς στα πλαίσια και της εργασίας σας και της εκθεσής σας, ή μάλλον καλύτερα για το θέμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε το Eurojust στην εργασία του. Να έχει τους αναγκαίους πόρους, τις δυνατότητες που του χρειάζονται για να λειτουργήσει το γραφείο του ε, εισαγγελέα. Και να ενισχύσουμε τα μέσα που έχουμε και αναπτύξει και αναπτύσσουμε με τη δική σας στήριξη για να υπάρξουν περισσότερες διαμεθοριακές ε, συνεργασίες. Για παράδειγμα, η, εντολή, η ευρωπαϊκή εντολή Έρευνα είναι πολύ σημαντική. Και οι προτάσεις ε, που έχουμε κάνει για την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία που χρειάζονται για περισσότερες ε, επιτυχείς διώξεις. Πολλά από τα στοιχεία αυτά είναι σε ηλεκτρονική μορφή και πολλές φορές ε, ανήκουν σε άλλη δικαιοδοσία. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες που να διευκολύνουν την πρόσβαση και τη συνεργασία. Ελπίζω λοιπόν να σημειωθεί ταχεία πρόοδος και σε αυτά τα θέματα. Αυτά είναι κάποια βραχυπρόθεσμα ζητήματα που ελπίζω ότι θα βοηθήσουν. Αν τώρα έχω κάπως ε, πιο μακροπρόθεσμη προοπτική Νομίζω ότι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων του γραφείου του Ισαγγελέα θα βοηθήσει να καταπολεμηθεί ο κατακαιρματισμός των ερευνών που αφορούν πολλές χώρες της Ένωσης για τόσο βασικά θέματα όπως είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και μαζί με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που ανέφερα και στα οποία νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε νομίζω ότι γενικά η μέσοπρόθεσμη προοπτική είναι θετική και χρήσιμη. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα οι σκιώδεις μας. Πρώτα απ' όλα η Κατερίνα Τσινίτσι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τον ε, Επίτροπο Κίνγκ που είχε την καλοσύνη σήμερα να έρθει στην Επιτροπή μας για να καταγράψει τις εξελίξεις, την τόση δουλειά που έχει γίνει και αν μου επιτρέπετε μια προσωπική παρατήρηση. Εμένα ως Ιταλίδα με χαροποιεί ιδιαίτερος που άρχισε μιλώντας για τον καφέ που πίνει. Πέραν αυτού, Σε ευχαριστώ πολύ και για τη δουλειά που προάγεται και για το γεγονός ότι έρχεστε και βέβαια να μας ενημερώσετε για τη δουλειά που κάνετε, αλλά και να μας ακούσετε και να ενημερωθείτε και για τα δικά μας βήματα προόδου. Αυτό ενισχύει την δική μας αποφασιστικότητα ε, στην προσπάθεια που κάνουμε για να προωθήσουμε το έργο μας. Ιδιαιτέρως ε, ορίζω τις πρωτοβουλίες, όλες τις πρωτοβουλίες για όλα τα νέα νομοθετήματα στα οποία αναφερθήκατε και τα οποία θα ε, παρουσιάσουν ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας. Ασφάλεια στην οποία κατά προτεραιότητα απαιτεί ο Ευρωπαίος πολίτης και βλέπουμε δυστυχώς ότι κάποια κράτη-μέλη καθυστερούν στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκών ε, διατάξεων και νομοθετημάτων που έχουν ακριβώς εισαχθεί προκειμένου να εξασφαλίσουν την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών και την αντιμετώπιση των ε, τρομοκρατικών επιθέσεων και απειλών. Και θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι μπορούμε στον κοινοβουλευτικό διάλογο να βρούμε μια καλή συμβαστική λύση και στο θέμα της διαλειτουργικότητας. Θέματος περιπλοκού, ναι, δύσκολου, ναι, που οπωσδήποτε όμως μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο προόδου και θα συμβάλλει αν τα καταφέρουμε να, ε, στην αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής. Ε, κατόπιν αυτών των εισαγωγικών λοιπόν παρατηρήσεων, θα αναφερθώ στις συγκεκριμένε ομοθέτικες προτάσεις ε, τις οποίες αναφέρατε και εσείς, αλλά κυρίως θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της προπαγάνδας μίσους και της διαδοσής της διαγραμμικά. Ε, είπατε ότι πρέπει μέσα σε μια ώρα να σβήνεται το σχετικό περιεχόμενο, να διαγράφει το σχετικό περιεχόμενο μίσους. Ε, θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι αυτή αυτή η μία ώρα, η διορία που λέτε ότι θα πρέπει να δίνεται για τη διαγραφή του περιεχομένου θα πρέπει να αφορά η αδίποτε επιχείρηση του τομέα. Θα μπορούν ενδεχομένω μικρότερε επιχειρήσει που άρα έχουν και, και λιγότερου πόρου διάθεσή του να έχουν μια κάποια προτεραιότητα τρόπον τι να μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Θεωρείτε ότι είναι δυνατόν μέσω αυτών των προτάσεων και των διατάξεων της πρότασης να προ, προληφθεί το ενδεχόμενο, όπως συχνά συμβαίνει, το περιεχόμενο που διαγράφεται από τη μια πλατφόρμα να αναφαίνεται σε μια άλλη και που τελικά ε, είναι το πρόβλημα. Και επίσης η Europol που έχει κάνει τόσο πολύ καλή δουλειά. Σε ποιο βαθμό συμβάλλει, με ποιο ρόλο μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την σηματοδότηση, τη σήμανση αυτού του περιεχομένου. Επίσης, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος για όλη την ε, ε, αντιμετώπιση και τα σχόλια που κάνατε για τα τροπολογίες μας είναι πάρα πολλές. Βέβαια δείχνει αυτό που είπατε κι εσείς πόση πολλή δουλειά κάνουμε κι εμείς ξέροντας ότι καθήκον έχουμε να συμβάλλουμε στο μέγιστο στον αγώνα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής. Και επίσης για να συμφωνήσω με τόσα επιναταλή ε, οπωσδήποτε πρέπει και στην προσεχή θητεία να, να παραμείνει ένα χαρτοφυλάκιο, μια θέση Επιτρόπου για τα θέματα της τρομοκρατίας ε, για να συνεχιστεί αυτή η καλή δουλειά. Επίσης, κάποια συγκεκριμένες παρατηρήσεις τώρα, αν μου επιτρέπετε. Ένα θέμα που μας αφορά και μας απασχολεί όλους είναι αυτό της προστασίας των θυμάτων και των οικείων. Τους ξέρετε ότι υπάρχει μια ε, πρόταση για τον συντονισμό της προστασίας των θυμάτων των επιθέσεων των τρομοκρατικών. Θα ήθελα να μου το σχολιάσετε και επίσης το θέμα της ιδιαίτερης προσοχής που πρέπει να δοθεί ώστε να μην υπάρχει σύγχυση στα θέματα, στην εικόνα σύγχυση σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές και την παρουσία τρομοκρατικής απειλής μέσω αυτών. Ε, και βέβαια πρέπει να κοιτάξουμε και τη ριζοσπαστικοποίηση που μπορεί να προκύπτει μέσα από τις φυλακές ή και έξω από αυτές. Αυτά αν μπορείτε να μου σχολιάσετε σε σχέση με τις προτάσεις ε, που έχουμε διατυπώσει μέσω των τροπολογιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και βέβαια ευχαριστώ και την Αταλή. Ευχαριστώ κύριε Σουπίτροπος. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Να επιχειρήσω να απαντήσω. Αλλά ίσως μπορεί κάποιες να τις ξανασυζητήσουμε και αργότερα πιο αναλυτικά αν χρειαστεί, αν υπάρχει ενδιαφέρον. Πρώτον, διαλειτουργικότητα. Όπως είπα και στην ομιλία Ναι, το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Και ελπίζω να βρούμε τρόπο να ολοκληρώσουμε την εργασία μας επ' αυτού. Ξέρω ότι το θέμα αυτό είναι επίμαχο, τους ανησυχεί ορισμένους. Αλλά κοιτάξτε, ας ε, δούμε λίγο το ευρύτερο πλαίσιο. Γιατί ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια. Διότι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή, οι αστυνομικοί, οι συνοριοφύλακες και άλλοι, αυτοί που η δουλειά τους είναι ακριβώς να μας διατηρούν ασφαλείς, μας είπανε όταν τους ρωτήσαμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Μας είπαν λοιπόν ότι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνεχώς είναι ότι το δίκτυο των ε, βάσεων δεδομένων που υπάρχουν στις διάφορες χώρες της Ένωσης είναι πολύ περίπλοκο, ε, πολύ γραφειοκρατικά διαμορφωμένο, δεν τους βοηθάει. Δεν είναι επειδή εγώ ή κάποιος από την Επιτροπή καθόμουν κάπου στο γραφείο μου και σκεφτόμουν τι μπορώ τώρα να προτείνω που γι' αυτό διατυπώθηκε αυτή η πρόταση. Μα το είπαν αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή τη μάχη. Μα είπαν ότι κάθε μέρα του δημιουργεί προβλήματα αυτή η κατάσταση. Εξετάσαμε λοιπόν τι τεχνικά μέτρα θα μπορούσαμε να πάρουμε. Μέσω των τεχνικών ε, της ε, τεχνολογίας, της πληροφορίας για να τους βοηθήσουμε. Και Αυτά που προτείνονται είναι τεχνικά, μπορεί να μην είναι πολύ συναρπαστικά όταν τα βλέπει κανείς, είναι πώς θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς τις δυνατότητες έρευνας για να λάβει πληροφορίες που ήδη υπάρχουν σε διάφορες τράπεζες ε, ή βάσεις δεδομένων ή και εκτός αυτών, όσο πιο γρήγορα γίνεται, με κάθε σεβασμό για τα, πολλά, ε, για τα πολύ υψηλά επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων. σε κάποιες συζητήσεις. Αυτό έχει γίνει τώρα κάτι που συνδέεται με άλλες ανησυχίες τους. Το κατανοώ. Αλλά θυμηθείτε από πού προέκυψαν αυτές οι προτάσεις και μελετήστε το ακριβές περιεχόμενό τους. Και, και σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και σε οποιοδήποτε πλαίσιο, είμαι απόλυτα διατεθειμένος να μπω σε κάθε τεχνική λεπτομέρεια, αν το επιθυμείτε, για να συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις. Γιατί δεν θεωρώ ότι ορισμένες από τις ανησυχίες που εκφράζονται είναι όντως βάσιμες. Για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, για το τι ίσως με κάποιο τρόπο αυτό να ανοίξει την πόρτα για εκτεταμένη ε, εξόριξη στοιχείων που μπορεί να ε, αποβεί ει βάρος ε, κάποιων κατηγοριών ε, ατόμων στην Ευρώπη. Καταλαβαίνω αυτές τις ανησυχίε. Αλλά δεν βλέπω πραγματικά να στοιχειοθετούνται από τις προτάσεις μας. Αυτά γενικά και είμαι απόλυτα διατεθειμένο να συζητήσω με όλους σας για το θέμα αυτό τώρα ή οποτεδήποτε άλλοτε θέλετε. Τώρα, άλλα θέματα. Οι προτάση μας ε, για να αντιμετωπίσουμε το παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο. Υπάρχουν διάφορα είδη επιβλαβούς ε, επιγραμμικού περιεχομένου. Και δεν λέμε ότι υπάρχει μία λύση για όλα αυτά τα είδη. Πολλά θέματα έχουν να κάνουν με τις ψευδείς ειδήσει, την παραπληροφόρηση. Και εκεί θα ε, διατυπώσουμε ένα κώδικα διοντολογίας και άλλα μέτρα δεν ε, ε, θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο να πούμε αν είναι αλήθεια ή όχι. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το κάνει, αλλά μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερη διαφάνεια για τις ε, πολιτικές συζητήσεις στο ίντερνετ, να ξέρουμε περισσότερο για από πού προέρχεται οποιοδήποτε υλικό αναρτάται και αυτό κάνουν και οι επίτροποι Γκάβριελ και Γιούροβα. Και μετά υπάρχουν κάποια είδη περιεχομένου που πρέπει να μας ανησυχούν. Για παράδειγμα, περιεχόμενο ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εκμετάλλευσης των παιδιών, όπου έχει υπάρξει ήδη νομοθεσία. Πώς ε, τα κράτη-μέλη θα αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα που ανεβαίνουν τέτοιο περιεχόμενο όταν αναρτάται στις πλατφόρμες. Τώρα θέλουμε να καταπολεμήσουμε το παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο. Υπάρχει σαφής ορισμός για το τι είναι τρομοκρατία. Δεν λέμε ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν για τα λεγόμενα κηρύγματα μίσους. Γιατί εδώ οι ορισμοί είναι ε, λιγότερο σαφείς. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι από χώρα σε χώρα, με βάση την ε, διαφορετική ιστορία, τις διαφορετικές παραδόσεις τους, έχουν διαφορετική προσέγγιση για διάφορα είδη κηρυγμάτων μίσους. Η Γερμανία αποφάσισε, για παράδειγμα, να προωθήσει νομοθέτημα, Άλλες όχι. Δεν υπάρχει ομοφωνία στο ευρωπαϊκό επίπεδο για τον ορισμό του, των κηρυγμάτων μίσους που να μας επιτρέψει να προωθήσουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αλλά για την τρομοκρατία έχουμε. Έχει συμφωνηθεί ένας ορισμός στην οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχουμε τους ορισμούς των Ηνωμένων Εθνών και νομίζω ότι μπορούμε ακριβώς να στοχεύσουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο για να πάρουμε στοχευμένα μέτρα. Αναφέρατε ένα μέτρο για τη μία ώρα. Ισχύει αυτό όταν κάποια αστυνομική ή δικαστική αρχή έχει εντοπίσει υλικό που θεωρεί ότι είναι παράνομο. Παράνομο, άρα παραβαίνει τον νόμο. Ενημερώνουν την πλατφόρμα, τη στέλνουν εντολή, την οποία πρέπει να εφαρμόσει μέσα σε μία ώρα. Αυτό βοηθάει νομίζω τις μικρές πλατφόρμες, γιατί αυτή τη στιγμή όλα είναι λίγο πιο φλού και οι πλατφόρμες εργάζονται με βάση τον όρο λειτουργίας τους και οι πλατφόρμες ε, έχουν πολύ προσωπικό που ασχολείται με αυτό, οι μεγάλες πλατφόρμες που έχουν πολύ προσωπικό που ασχολείται με αυτό, έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες να αντιδράσουν ε, από ό,τι έχουν οι μικρότερες πλατφόρμες. Με αυτό τους λέμε, δεν σας ζητάμε να κρίνετε αν αυτό το περιεχόμενο ανταποκρίνεται στους όρους λειτουργίας σας, αν σας αρέσει, σας λέμε ότι είναι παράνομο το περιεχόμενο και οι αρχές σας ενημερώνουν ότι είναι παράνομο και να το βγάλετε. Εκτελέστε την εντολή που λάβατε. Φυσικά, από πίσω πρέπει να έχουμε πολύ ρωμαλές ασφαλιστικές δικλείδες και εγγύησεις. Και αυτές που προτείνουμε και που θα τις συζητήσουμε αναλυτικότερα και με εσάς, είναι ιδιαίτερος ρωμαλές, πιο ρωμαλές, πιο πλήρης από ό,τι υπάρχει τώρα. Υπάρχει υποχρέωση διαφάνειας, θα πρέπει να αναγγείλουν ποιο υλικό κατεβάζουν και υπάρχουν και μηχανισμοί προσφυγής και υπάρχει και δυνατότητα δικαστικής προσφυγής. Αν λοιπόν κάτι λανθασμένα αφαιρεθεί, μπορεί κανείς να προσφύγει. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφιβάλλω ότι δεν είναι επαρκώς διαφανές κάτι τέτοιο και δεν θεωρώ ότι πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις θα υποβάλουν ε, παράπονα προσφυγές. Αλλά αν γίνει κάποιο λάθος και αν κάποιος ε, προσφύγει, το υλικό έχει παραμείνει και μπορεί να επαναναρτηθεί. Η Europol πρέπει να συνεχίσει να παίζει βασικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουν ένα ειδικό όργανο, το IRU, και θέλω να χαιρετήσω την εργασία που κάνουν και νομίζω ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει να μας δίνει η Europol την εμπειρογνωμοσύνη της σε όλα τα κράτη-μέλη όσο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Για τα θύματα, ε, ε, να επανέλθω όταν γίνουν άλλε ερωτήσει, Φυσικά είναι βασική προτεραιότητά μας. Έχουν γίνει διάφορα βήματα. Νομίζω ότι ε, είχα παρουσιάσει και εδώ ε, τα θέματα αυτά και φυσικά θα συνεχιστούν τα πιλωτικά προγράμματα και όπως είπα το πρώτο βήμα είναι τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την αντιτρομοκρατική οδηγία που περιέχει και ε, διατάξεις για τα θύματα για την ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές, ε, να επανέλθω εάν το θέλετε περισσότερο. Είναι βασικό ζήτημα που έχει προκύψει από την εργασία που έχουμε κάνει το τελευταίο χρόνο στην ε, ομάδα υψηλού επίπεδου για την αντιμετώπιση της ε, ριζοσπαστικοποίησης, όπου είχαμε εμπειρογνώμονες όχι μόνο από την κοινωνία των πολιτών, αλλά και από τη δημόσια διοίκηση και από την κεντρική διοίκηση για να συγκρίνουμε τις εμπειρίες μας. Κανείς δεν εκπλήσεται που οι φυλακές είναι μια βασική προτεραιότητα. Σήμερα το πρωί διάβασα στις ειδήσει ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, τονίζεται η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές. Θα είναι μία από τις προτεραιότητές μας στις συναντήσεις που θα έχουμε όταν ξεκινήσει μάλιστα η νέα πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης κατά τη διάρκεια του μηνός. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Δίνετε σαφέστατες διευκρινήσεις και κάπως έτσι διευκολύνεται τα πράγματα. Αλλά για το θέμα της διαλειτουργικότητας θα χρειαστεί να κινητοποιήσουμε όλοι μας την πυθό ε, προς τους συναδέλφους. Το λόγο κυρία Μάιτε Παγκασαουρτουντούα. Επίσης και οδησηγήτρια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που όπως πάντα δίνει διαφανείς πληροφορίες ε, και είναι πολύ προσινής. Μιλήσατε για το θέμα της Ισπανίας και τη ριζοσπαστικοποίηση στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Αν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία, στι 40% των περιπτώσεων ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές της Ισπανίας έχουν σχέση με άτομα που έχουν ήδη προηγούμενη ριζοσπαστικοποίηση συμπεριφορά Δεν είναι ιδεολογική. Πρόκειται για άτομα που ήδη έχουν ένα εγκληματικό παρελθόν και είναι πολύ πιο πρόσφορα, πιο επιρρεπή στη ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές. Τουλάχιστον στην Ισπανία αυτό παρατηρήσαμε και είναι πολύ σημαντικό το φαινόμενο και θα πρέπει να προσδιορίσουμε πώς, ε, αν κάποιος έχει ήδη ριζοσπαστικοποιηθεί και έχει καταδικαστεί για τρομοκρατικά εγκλήματα, μπορεί να προσελκύσει και κοινού εγκληματίε. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε πολύ ρεαλιστικά. Κύριε Επιτροπέ, μιλήσατε για την αφαίρεση διαγραφή περιεχομένου μετά από αστυνομικό ή δικαστικό ένταλμα. Θα ήθελα αυτό να μας παρουσιάσετε, γιατί δεν είναι το ίδιο ένα ένταλμα αστυνομικό με ένταλμα που έχει εκδοθεί από δικαστή. Δεν είναι δηλαδή το ίδιο ένα μέτρο δικαστικού ελέγχου με ένα διοικητικό μέτρο. Από τις εξηγήσεις που μας δώσατε καταλάβαμε ότι μία ώρα διορία για τις τεχνολογικές πλατφόρμες είναι σημαντικός χρόνος. Κάτι που σημαίνει ότι προηγουμένως είχαμε έκθεση σε αυτό το περιεχόμενο που κρίθηκε παράνομο. Το θέμα του δικαστικού ελέγχου με ενδιαφέρει ιδιαίτερος, γιατί όταν γίνονται επεμβάσεις ε, σε στοιχεία, σε δεδομένα ή σε προσωπικές ανακοινώσεις ή μηνύματα, ε, πριν το διαδίκτυο, το θέμα του δικαστικού ελέγχου είχε θεμελιώδη σημασία. Πριν από 30-40 χρόνια, είχαμε την επέμβαση στα τηλέφωνα που γινόταν χειροκίνητα μετά από το δικαστικό ένταλμα. Ε, γινόταν, ε, έπρεπε να δοθεί δικαστικό ένταλμα για επέμβαση στα, τηλεφωνικά μηνύματα. Εδώ όμως έχουμε ένα τεράστιο φάσμα δυνατότητας ε, επέμβαση στα δεδομένα ή στα προσωπικά μηνύματα. Πώς θα εξασφαλίσουμε τα ειχέγγυα. Και όταν μιλήσατε για την αντιτρομοκρατική οδηγία, αυτή οδηγία σίγουρα είναι σημαντικότατο εργαλείο και ήδη από το Σεπτέμβριο έχει, έπρεπε να είχε μετατεθεί στην εσωτερική ενόμη τάξη, οπότε πολύ πρόσφατα. Και είπατε ε, μόνο πέντε χώρες την έχουν εφαρμόσει μέχρι στιγμής. Τι εννοείτε, δηλαδή ότι τυπικά την έχουμε μεταθέσει στην ένωμη του τάξη ή ήδη ελέγξατε αν από άποψη περιεχομένου εφαρμόζουν ήδη την οδηγία αυτές οι πέντε χώρες. Τι ακριβώς εννοούσατε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και είναι και σημαντικότατο εργαλείο αυτή η οδηγία και με σωστή ενημέρωση θα μπορέσουμε και εμείς να επηρεάσουμε τα πράγματα. Και είπατε όταν δεν θα είστε πια επίτροπος θα δούμε. Σας ευχαριστώ, Μάιτε. Μία μικρή προσθήκη, ένα συμπλήρωμα στην ερώτηση της Μάιτε για τις χώρες που έχουν ε, εμπρόθεσμα μεταθέσει την ε, οδηγία στην εσωτερική του ένωμη τάξη. σω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ρόλο θα παίξετε, μια και είστε θεματοφύλακα των συνθήκων. Πινκ-πονγκ έχουμε, οπότε ε, θα απαντήσετε. Ναι, πραγματικά δεν έχω κι εγώ ιδέα ποιο θα ακολουθήσει, αλλά ελπίζω κάποιο να με διαδεχθεί. Αυτό είναι το βασικό, κάποιο να αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις με αντίστροφη σειρά από αυτή που τις θέσατε. Στην έκθεση της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε διεξοδικές ε, πληροφορίες ε, ανά νομοθετικό εργαλείο, ε, τι γίνεται με τις κοινοποίησεις σε που έχουμε τις επίσημες κοινοποίησεις. Και αυτό που μας εντυπωσιάζει με την οδηγία για την αντιτρομοκρατία. Και ήταν εντυπωσιακό ότι ήταν πολύ σημαντική οδηγία, προβλήθηκε ιδιαίτερο και δώσαμε και τη διορία για την κοινοποίηση. Όταν όμως τον περασμένο μήνα έληξε η διορία, μόνο πέντε χώρες επίσημα κοινοποίησαν τη μεταγραφή. Ελπίζουμε, και αυτό το ερευνούμε τώρα, το διερευνούμε, ότι και άλλες χώρες ε, μέλη έχουν προχωρήσει στη θέσπιση μέτρων που προβλέπει η οδηγία για την αντιτρομοκρατία γιατί πολύ συχνά υπάρχει μια χρονική υστέρηση μεταξύ της ε, θέσπισης των μέτρων και της επίσημης κοινοποίηση. Οπότε ελπίζω ότι το πήρουν είναι κάπως καλύτερο, κάπως πιο ελπιδοφόρο. Πάντως ε, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί η οδηγία για την αντιτρομοκρατία είναι πολύ σημαντική και θέλουμε να εφαρμοστεί. Θέλουμε ο αριθμός των χωρών που ε, επίσημα κοινοποίησαν την εφαρμογή να αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά και ταχαίως. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας για τη διορία της μίας ώρας για την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου που έχει σχέση με την τρομοκρατία. Τα κράτη-μέλη, με βάση την νομοθεσία τους, έχουν αρμόδιους φορείς και αρχές που μπορούν να εκδώσουν το ένταλμα αφαίρεση ή διαγραφή περιεχομένου. Και θα πρέπει στι ασφαλιστικέ δικλείδε που προτείνουμε να είμαστε σαφεί αν πρόκειται για προσφυγή ή ερώτηση είτε από την ε, λόγω πλατφόρμα ή από τον συντάκτη του περιεχομένου, σε περίπτωση που αφαιρεθεί το περιεχομένο και ενημερωθεί, τα ένδικα μέσα θα πρέπει να είναι πραγματικά ένδικα, δικαστικές προσφυγές. Οπότε προσπαθούμε έτσι να εξισορροπήσουμε την ανάγκη ταχεία αντίδρασης, γιατί αν αφήσουμε το περιεχόμενο στην πλατφόρμα θα διαδοθεί, θα εξαπλωθεί και να το συνδυάσουμε αυτό και να το συμβάσουμε με την ανάγκη να έχουμε μία δικαστική διαδικασία άσκησης προσφυγών ή ένδικων μέσων. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή την πιθανότητα δικαστικού ελέγχου. Σε ό,τι αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές, συμφωνώ ε, πολύ εύστοχα και εύγλωτα μιλήσατε για το πρόβλημα που έχουμε με το ακροατήριο που προσελκύεται, γιατί δεν είναι όλοι οι ριζοσπαστικοποιημένοι στις φυλακές ε, άνθρωποι που πήγαν στις φυλακές ε, για ιδεολογικούς λόγους και ριζοσπαστικοποιήθηκαν για ιδεολογικούς λόγους ή φυλακίστηκαν για τρομοκρατικές ενέργειες. Πολύ συχνά αυτοί που στρατολογούνται και ριζοσπαστικοποιούν τις φυλακές φυλακίστηκαν για άσχετους λόγους, είναι κοινοί εγκληματίες. Και όπως είπατε είναι υψηλό το ποσοστό των περιστάσεων που μερικές φορές ανήλικοι ή άσχετοι με την τρομοκρατία, ή άσχετοι με την τρομοκρατία εγκλήματα φυλακίστηκαν. Βέβαια δεν είναι ανήλικοι γιατί όντως έχουν φυλακιστεί. πάντως φυλακίστηκαν ή καταδικάστηκαν για εγκλήματα άσχετα με την τρομοκρατία. Και στις φυλακές ριζοσπαστικοποιήθηκαν από δίκτυα τρομοκρατών που στρατολογούν τρομοκράτες. Βέβαια δεν υπάρχει καμία μαγική λύση και τα κράτη-μέλη με διαφορετικούς τρόπους το χειρίζονται και προσπαθούν να το λύσουν. Άλλοι ομαδικά ε, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους ροζοσπαστικοποιημένους, άλλοι προσπαθούν να τους διαχωρίσουν, να τους μοιράσουν. Ε, κάθε κράτος χρησιμοποιεί τη δική του προσέγγιση. Θα συγκεντρώσουμε αυτές τις προσεγγίσεις και του χρόνου θα σας ενημερώσουμε και εσάς και όσους παρακολουθούν το θέμα, έχοντας μια ανοιχτή συζήτηση για τα διδάγματα που αντλήσαμε από τις διάφορες εθνικές εμπειρίες. Και όπως ξέρετε, χρηματοδοτούμε πολλά προγράμματα για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές. Και θα δούμε αν χρησιμοποιείται χρηματοδότηση αποτελεσματικά ή χρειάζεται συμπλήρωσή της. Πάντως, το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διδαχθούμε από τις εμπειρίες των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Je passe la parole. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην αντιπρόεδρο μα τώρα, την κυρία Βαλενσιάνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και τον Επίτροπο για την παρουσία του, για το έργο του που θα παραμείνει για το μέλλον, άσχετα με το ποιος θα είναι ο διάδοχός σας και άσχετα με το ποιο θα είναι το επόμενο κοινοβούλιο μετά τι ευρωεκλογέ, γιατί ούτε και εμεί γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι δικοί μα διάδοχοι και αν θα συνεχίσουμε εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντω, κάτι που με προβληματίζει πρόσφατα και έχει σχέση με την παρουσία ε, στο δημόσιο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η αντίδραση των ευρωπαϊκών κοινωνιών είναι πάντα μια άμεση αντίδραση θερμό, μετά από μια καταστροφή, μετά από μια τρομοκρατική απόπειρα, τότε είναι που αυξάνεται κατακόρυφα η ευαισθησία του κοινού. Αλλά στο μέτρο που δεν έχουμε τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις, παρόλο που υπάρχουν σε άλλα μέρη του κόσμου τέτοιες και συνεχίζονται, από τη στιγμή που δεν μας αγγίζει άμεσα, η ευαισθησία του ευρωπαϊκού κοινού μειώνεται ε, και εξαφανίζεται το θέμα της αντιτρομοκρατίας από το πρόγραμμα το πολιτικό. Και αυτό είναι πολύ κακό, πολύ αρνητικό, γιατί θέλουμε αμύωτη την πίεση προς τα κράτη-μέλη για να μεταφέρουν τις οδηγίες στο εσωτερικό τους δίκαιο και να εξασφαλίζουν ένα συντονισμό μεταξύ τους. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι η τρομοκρατία είναι πολύ δυσάρεστο θέμα για ένα πολιτικό πρόγραμμα και σίγουρα οι πολιτικοί σε εθνικό επίπεδο, ε, αν μπορούν να το αναφέρουν, ε, να το παραλείπουν τόσο το καλύτερο. Το θέμα όμως είναι ότι η τρομοκρατία είναι παρούσα και Ασχολούμαστε με αυτή μόνο όταν μας επηρεάζει άμεσα, όταν μας αγγίζει. Οπότε το πολιτικό πρόγραμμα των κυβερνήσεων και εκεί ε, χαλαρώνουν όταν μειώνεται και η κοινωνική ευαισθησία σε περίπτωση που δεν υπάρχουν φαινόμενα τρομοκρατίας άμεσα. Αλλά είναι αναφυσβήτητο ότι τα βήματα θα τα πραγματοποιήσουμε μόνο αν προχωρήσουμε και κρατήσουμε αμοιότητη την πίεση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, 100%, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει. Ε, είναι αναγκαίο να ξεφύγουμε από την ε, προσέγγιση ε, την κατακαιρματισμένη, το σταματούμε και προχωρούμε. Αν έχουν περάσει 15-20 χρόνια από τη τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους Πολύ συχνά δεν είχαμε μία αμύωτη πίεση ή μία συνεχή διαδικασία, αλλά συνέχεια σταματάμε, προχωράμε, σταματάμε, προχωράμε. Και εδώ δύο είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. Τον πρώτο τον επισημάνατε. Για να είμαστε αποτελεσματικοί χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση και συνεχή. Ο δεύτερος κίνδυνος που προέκυψε από τη συζήτηση και είναι επίση σημαντικό: είναι ότι αν συνέχεια απλώς αντιδρούμε εν θερμό, αμέσως δηλαδή μετά μια τραγωδία, μια τρομοκρατική επίθεση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να κάνουμε λάθη στην ε, παρορμητική αντίδραση, στην εφερμό αντίδραση. Οπότε, όχι μόνο χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμη δέσμευση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, θα πρέπει να έχουμε και μακροπρόθεσμες προοπτικές κατά τη χάραξη των πολιτικών όσο και είναι πιο ικανοποιητικό να κάνουμε κάτι δραματικό άμεσα ε, την επαύριο τη τρομοκρατική επίθεση. Αλλά ίσω μια τέτοια θερμό αντίδραση δεν είναι η καλύτερη αντίδραση υπό πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Οπότε θα πρέπει να σταματήσουμε αυτό το φαύλο κύκλο. Σταματάμε, προχωράμε και δεν υπάρχει μια συνέχεια. Και πραγματικά το έργο σα ε, εμπίπτει σε αυτή την προσέγγιση τη ε, χάραξη μακροπρόθεσμη προοπτική και τη εμβριθούς ενασχόληση με το θέμα και τη συνεχού. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Να έχουμε δηλαδή συγκεκριμένου πόρου για τα θέματα τη ασφάλεια, συνδυάζοντα του διάφορου άξονε δραστηριοτήτων και υιοθετώντα μια μακρόπνοη, μακροπρόθεσμη προοπτική. Και συμφωνώ μαζί σα ότι θα πρέπει να συνεχίζουμε τις, ε, τα διαβήματά μας και προς τα κράτη-μέλη και με τις αρμόδιες αρχές και να υπάρχει αυτή η συνέχεια. Γιατί θα πρέπει αφού περνάει μια νομοθεσία, θεσπίζεται να θεωρούμε ότι λύθηκε το πρόβλημα. Γιατί όντω δεν λύεται μόνο με την νομοθεσία. Πρέπει πρώτα να εφαρμόζεται η νομοθεσία και μετά συνεχώς σταδιακά να επανερχόμαστε και επανειλημμένως να επανερχόμαστε στα θέματα και να μην τα ξεχνούμε. Μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Επίσης, δεν θα πρέπει όλες αυτές τις προκλήσεις να τις αντιμετωπίζουμε μόνο υπό την ευρωπαϊκή σκοπιά. Θα πρέπει να τη δούμε και με το θέμα του, με βάση τον αντίκτυπο που έχει και στις κοινωνίες μας, στις πατρίδες μας, στις χώρες μας, αλλά υπάρχει άρρηκτος δεσμός μεταξύ αυτών των προβλημάτων. Είναι αλληλένδετα αυτά τα προβλήματα. Αυτά που συμβαίνει στους δρόμους μας και αυτό που συμβαίνει στη γειτονία μας και πιο μακριά είναι αλληλένδετα θέματα. Όσο μακριά και αν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, έχουν μια σύνδεση μεταξύ τους. Και αυτό το έχουμε και στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ΕΕΔ. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις γειτονικέ μας χώρες ε, και τους εταίρους μας διατλαντικά και αλλού να αντιμετωπίσουν την, την αντιτρομοκρατία και τη ριζοσ... την τρομοκρατία μάλλον και τη ριζοσπαστικοποίηση. Και πριν από 3-4 χρόνια καταφέραμε και είμαι περήφανος γι' αυτό ότι κινητοποίησαμε 2 δισεκατομμύρια ε, ευρώ βοήθεια προς τους γειτονές μας και τους εταίρους μας διατελετικά για να τους βοηθήσουμε, όχι διατελετικά, μάλλον γενικώ, να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία και να κινητοποιήσουν τις δυνάμεις τους. Θα πρέπει να δούμε και το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό προβληματίζει σίγουρα και εσά, αλλά περισσότερο ίσως άλλες επιτροπές είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικέ και να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση, όχι μόνο για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός, στα εξωτερικά μας σύνορα, αλλά και ε, να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας ε, και στο εξωτερικό με τους εταίρους ε, και γειτονέ μα. Ευχαριστώ πολύ, Σερ Τζούλιαν, και πριν να δώσω το λόγο στου τρει τελευταίου ομιλητέ μα και σημειώνοντα ότι έχουμε τήρηση τους χρόνους μας, διατηρώντας τη ρευστότητα της συζήτησης, χωρίς να πιέζουμε τους ομιλητές. Θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση της Ελένα, που είναι πολιτική, νομική, δημοσιονομικού χαρακτήρα, αλλά και κοινωνιολογικού. Θα σημειώσω. Μια μήνυ ερώτηση. Εσείς που διαρκώς έχετε επικοινωνία με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και ξέροντας ότι κράτη που έχουν ε, λίγο πολύ ε, πέσει θύματα τρομοκρατικών υποθέσεων, ε, έχουν δει τις συνέπειες. Εγώ ως Γαλλίδα βλέπω ότι ζω σε μια κοινωνία που υπάρχει ταυτόχρονα αυτό το παιχνίδι της απειλής και της αντοχής διαρκώς μέσα στους δρόμους μας, στους σταθμούς, στα καφενεία και ταυτόχρονα, ενώ υπάρχει απειλή λοιπόν πάντα παρούσα, έχουμε και την ε, ε, αντοχή, την ανθεκτικότητα, όντας μια κοινωνία τραυματισμένη από την απειλή και τις επιθέσεις. Εσείς βλέπετε κάποια αλλαγή νοοτροπία σε επίπεδο κυβερνήσεων, ε, των κρατών που δεν έχουν πληγεί από τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά που ενδεχομένως αισθάνονται πώς ε, οφείλουν να επιδείξουν αλληλεγγύη και να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε για να μην κερδίσουν οι τρομοκράτες αυτή την ε, αντιπαράθεση. Θα δώσω μετά το λόγο στους αδέλφους. Δεν είσαστε υποχρεωμένος να απαντήσετε φυσικά, αλλά είναι ένα γενικό το ερώτημα αυτό το οποίο με απασχολεί και μετά θα δώσω το λόγο στην Τερέζα Χιμένες. Όχι, ευχαρίστω να απαντήσω. Ή να σας μεταφέρω τις εμπειρίες μου γιατί δεν ξέρω αν θα είναι υπαρκής απάντηση. Ε, θα σας πω ότι διαισθάνομαι ε, σε επίπεδο όλων των κρατών μελών όλο και μεγαλύτερη σημασία να αποδίδεται στα θέματα της ασφάλειας. Βλέπω να μετατοπίζονται ίσως διαφορετικά οι προτεραιότητες ανάλογα το κράτος μέλος, αλλά πάντως εστιάζουν περισσότερο στο φάσμα των προκλήσεων των σχετικών με την ασφάλεια που έχουμε, σε σχέση με τις αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η καθημερινή μας ζωή, στον τρόπο διαβίωσης. Άρα βλέπουν μια σειρά από ε, προκλήσεις σχετικές με την ασφάλεια. Είτε είναι αυτές οι απειλές, η τρομοκρατία, είτε είναι οι κυβερνοεπιθέσεις των τελευταίων δύο ετών, είτε πρόκειται για πολιτική χειραγώγηση μέσω των, ε, της, ε, του, διαδικτύου, του κυβέρνου χώρου, που πάλι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μια ευαισθητοποίηση. Και επίσης βλέπω ότι τις απειλές αυτές τις ε, διαγιγνώσκουν είτε ως απειλές έξωθεν από άλλες χώρες ή κοινότητες, είτε ως προκλήσεις, όπως είπα, για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε τις αξίες ή τις συνθήκες διαβίωσης. Και γι' αυτό το λόγο ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις εστιάζονται σε αυτές τις προκλήσεις και θέλουν να συνδυάσουν τις απαντήσεις και την ανταπόκρισή τους. Και γι' αυτό το λόγο ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν την πρόταση και ιδέα για περισσότερες ε, και πιο συλλογικές προτάσεις και ε, ε, μέτρα αντιμετώπισης. Μερικέ φορέ μπορεί να προβάλλεται η έννοια τη επικουρικότητα, ω προ το ποιο θα κάνει τι ή πώ. Αλλά ε, αυτό όχι στον τομέα που με απασχολεί και στο δικό μου τομέα και πιστεύω θα με επιβεβαιώσετε κι εσείς, γιατί σε όλες τις επαφέ που έχω με τις κυβερνήσεις βλέπω ότι ενώ οι εθνικές αρχές, ε, κυβερνήσεις αναπόφευκτα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όταν τίθεται ζήτημα ασφάλεια των πολιτών τους, γιατί πρόκειται για τον πυρήνα των ε, ε, το, τον πυρήνα του πεδίου αρμοδιότητα μιας κυβέρνησης πάλι είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε όλο και πιο στενή συνεργασία γιατί ορισμού οι προκλήσεις αυτές ξεπερνούν τα σύνορα τα εθνικά μιας κοινωνίας, μιας κοινότητας, μιας κυβέρνησης και γι' αυτό βλέπουν ότι υπάρχει και μάλιστα και τη ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και βλέπουν ότι υπάρχει πάντα ανάγκη για μια προσέγγιση με εξωτερικό, προς το εξωτερικό στραμμένο το βλέμμα. Και γι' αυτό θέλουν να υπάρχει αυτός ο συντονισμός πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη για την ε, προστασία της ασφάλειας των πολιτών τους. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις, τις συζητούμε και εδώ. Προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση της εφαρμογής, αλλά στο, στις προθέσεις συμφωνούν τα κράτη. Ευχαριστώ Τερέσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την αποφασιστικότητά του, για την σαφήνειά του. και για το ενδιαφέρον του για τα θύματα. Ευχαριστώ και την κυρία Βαλεντιάνο που αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα εγώ είμαι και 9 χρόνια εδώ και βλέπω πώς ε, λειτουργεί η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και ξέρω πολύ καλά ότι βεβαίως ε, μόνο όταν, υπάρχει, όταν υπάρχουν έντονα συναισθήματα μετά από μια τρομοκρατική απόπειρα τότε προωθούμε κάτι τέτοια θέματα. Αυτό σημαίνει πως δεν γίνεται αρκετή προληπτική εργασία. Όλα γίνονται εκ των υστέρων. Όταν λοιπόν ε, δεν προσέχουμε αρκετά, τότε τους κάνουμε ακριβώς δώρα. Δεν πρέπει λοιπόν να επιτρέπουμε μέσω της έλλειψης ε, επαγρύπνησης να εποφελούνται. Θέλω να τονίσω ότι όπως είπε σωστά και η Ναταλή, και λένε ότι το γεγονό ότι δεν έχουμε τελευταία τρομοκρατικέ επιθέσεις δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή, σοβαρή έκθεση. Πήγαμε σε αεροδρόμια, μιλήσαμε με δικαστές, με αστυνομικού. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν μια πολύ σοβαρή έκθεση, όχι ιδεολογικού περιεχομένου. Θέλουμε να αναφέρουμε τις συγκεκριμένες τρομοκρατικές επιθέσεις όπως ε, το Ισλαμικό κράτος και πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε, διότι πρόκειται για την τρομοκρατία που είναι τόσο σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ορισμένε πολιτικέ ομάδε θέλουν να μην είμαστε σαφεί, δεν το καταλαβαίνω. Ίσως για ιδεολογικού λόγους, που δεν μας βοηθάει κάτι τέτοιο για να εργαστούμε αποτελεσματικά για την ασφαλεία μα. Μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα ε, τρομοκρατία και μετανάστευση χωρίς να λέμε ότι ε, το ένα είναι το ίδιο με το άλλο. Όχι, πρέπει να δούμε τι σχέση έχουν. Όταν μιλάμε για τις φυλακές, ε, επίσης το κάνουμε με τρόπο σοβαρό. Και πρέπει να είμαστε σοβαροί και βεβαίως πρέπει να ασχοληθούμε και με τα θύματα. Με ανησυχεί αυτό το οποίο είπατε για το ότι ορισμένοι εξυμνούν την τρομοκρατία. Βεβαίω δεν έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά θέλω να με εξηγήσετε τι ακριβώ εννοείτε. Και ποιοι ακριβώς ε, εξυμνούν την τρομοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στη χώρα μου για τα θύματα. Και υπόθηκε ότι πρέπει να υπάρχει μια υποεπιτροπή ε, μόνιμη για θέματα ασφάλειας που θα βοηθούσε να προωθήσουμε τα θέματα αυτά. Γιατί προς στιγμή δεν προωθούνται όσο θα έπρεπε δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή, γιατί είναι απρόθυμα τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Μόνο ενεργούν όταν ε, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, όταν ακριβώς έχει εστιάσει η κοινή γνώμη σε κάποια τέτοια θέματα. Και επιπλέον, τι νομίζετε εσείς ότι πρέπει να γίνεται με, τις, ε, με τα εντάλματα έκδοσης ε, που δεν εκτελούνται. Έχουμε ε, ένα ένταλμα έκδοσης για κάποιον που δεν έχει που δεν έχει ακόμη εκδοθεί, έχουν αποκαλυφθεί και άλλα πολύ σοβαρά εγκλήματά του, έχει ζητηθεί από την Ισπανία να εκδοθεί στο Βέλγιο, αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει μια ελάχιστη δικαστική συνεργασία. Δεν υπάρχει αυτή η δικαστική αρρωγή μεταξύ κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αν μου επιτρέπει ο Επίτροπος, θα δώσω λόγο και στην Χριστίνα Βίνμπεργκ και μετά στον Τόρου Φρουντζούλικα και μετά ε, να απαντήσετε συνολικά για να σεβαστούμε το χρόνο μας. Χριστίνα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσία του είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον να σας ακούμε. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ως ένα εγχείρημα για να υπάρξει ειρήνη, για να εγγυηθούμε την ειρήνη και την ασφάλεια στους συμπολίτες μας και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαζόμεθα, ιδίω σε περιόδους όπως αυτές που ζούμε τώρα. Όπως και προηγουμένως η Χέλγια Στίβενς έθεσε κάποια ερωτήματα που και εγώ ήθελα να θέσω. Για παράδειγμα, πώς εφαρμόζονται διάφορες οδηγίες, για παράδειγμα το PNR. Είπαμε ότι θα πρέπει μέχρι τον, ε, την άνοιξη του 18 το αργότερο να έχει υπάρξει πλήρης εφαρμογή. Όμως αυτό δεν έχει ε, ε, καταστεί πραγματικότητα. Αυτό μου φαίνεται εντελώ παράλογο. Έχουμε τόσες οδηγίες και όμως δεν εφαρμόζονται και η ριζοσπαστικοποίηση είναι απόλυτα ζωτική σημασία. Εδώ πολύ συχνά αναφερόμεθα στο ίντερνετ. Πώ μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την προπαγάνδα μέσω του ίντερνετ και νομίζω ότι έχουμε σημειώσει επαρκή πρόοδο. Αλλά οι φυλακέ είναι ένα άλλο θέμα που μα απασχολεί. Και οι φυλακέ πρέπει να είναι στο επίκεντρο τη προσοχή. μας. Μόλι διάβαζα στα γαλλικά μέσα ότι περίπου 40 άτομα έχουν καταδικαστεί για, που έχουν καταδικαστεί για τζιχαντιστικά εγκλήματα θα απελευθερωθούν. Και ένας Γάλλος εισαγγελέα λέει ότι η ριζοσπαστικοποίηση εντός των φυλακών είναι εντονότερη τώρα παρά ποτέ ε, στο παρελθόν. Και κάτι άλλο που δεν ε, συζητάμε πολύ συχνά ίσως είναι κάποια κράτη-μέλη απέτυχαν στις προσπάθειες να ενταχθούν ε, οι μειονότητες στη χώρα τους. Ε, ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα που διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές περιθωριοποιημένες ε, γειτονιές όπου οι έφηβοι και τα παιδιά ζουν σε εγκληματικό περιβάλλον, ε, ακούγονται πυροβολισμού, πυροβολισμοί κάθε δεύτερη μέρα, αυτοκίνητα καίγονται και ο Σουηδός Ομπούτσμαν έχει τονίσει ότι υπάρχουν ολόκληρες τέτοιες περιοχές όπου υπάρχει έντονη ριζοσπαστικοποίηση. Γιατί αυτοί οι νέοι ζουν σε κατάσταση χωρίς διέξοδο. Η κατάστασή τους είναι απεγνωσμένη. Και η Σουηδία ξέρουμε ότι εξάγει τρομοκράτες σε πολλέ άλλες χώρες μέλη. Οπότε γίνεται πρόβλημα και για εσά. Πώς αντιμετωπίζετε τι κατάσταση; Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φρουτζούλητσα, ζητώ συγγνώμη μου που έφτασα με τόση καθυστέρηση, αλλά έχουμε ταυτόχρονα πολλέ συνεδριάσει. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Τρεις πρακτικές ερωτήσεις. Καταρχάς, ε, θεωρείτε ότι χρειάζεται νέα νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, πρόληψη και την πάταξη της τρομοκρατίας. Δεύτερον, βεβαίως τα θέματα της ασφάλειας ε, παραμένουν αρμοδιότητα των κρατών μελών κατά κύριο λόγο. Ωστόσο, θεωρείτε ή πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα να ζητήσει από τα κράτη-μέλη την διάθεση περισσότερων πόρων για την πάταξη της τρομοκρατίας, ε, υλικών, οικονομικών, ε, ανθρώπινων, τεχνικών και άλλων πόρων για τις ορισμένες χώρες είναι πολύ κακή η κατάσταση και είναι ε, σε αδυναμία να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατική απειλή. Το ξέρετε αυτό. Και τρίτον, πώς μπορούν να παρακολουθούν ακολουθούνται και να εξασφαλιστεί μια ενό είδου τυποποίηση για τις βάσεις δεδομένων, γιατί ξέρετε πάντα αυτό είναι το πρόβλημα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα για πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τόσες βάσεις δεδομένων και δεν μιλώ για Σέγγεν και Προυμ και όλα τα άλλα που είναι μεταξύ τους ε, άσχετες, δεν υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα και γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να βελτιωθεί για να αντιμετωπίσουμε τη δημοκρατία. Κύριο Χιλ, έχετε το λόγο για όλη αυτή την ε, πληθώρα ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα και στην αρχή, επαναλαμβάνω κλείνοντας ότι σας ευχαριστώ θερμά για την προσήλωση στην αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων, τη δουλειά σας στην Επιτροπή και ιδιαίτερα το σχέδιο έκθεσης. Θεωρώ ότι η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική. Για τους λόγους που η κυρία Χιμένες, όπως και άλλοι, ιδιαίτερα υπογράμμισε. Μιλούμε για μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τα θέματα αυτά, που οπωσδήποτε θα πρέπει να στηρίζεται σε πρακτικά μελήματα, αλλά και επιπλέον αν μου επιτρέπετε τοποθέτηση, δεν θα πρέπει να προχωρεί με βάση βραχυπρόθεσμους μόνο σχεδιασμούς. Χρειάζεται μακροπρόθεσμη θεώρηση για να οριστούν ε, και όπως είπα και τα πλαίσια πάνω, μέσα στα οποία θα κινηθούν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσοχής αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσείς θα πρέπει να τα προσδιορίσετε αυτά τα πλαίσια και τα χρονοδιαγράμματα και ελπίζω να είσαστε φιλόδοξοι σε αυτό το στόχο. Επίσης συμφωνώ ότι πρέπει να δείξουμε προσοχή να μην ε, σφαλίσουμε τα θέματα ε, είτε είναι η κυβερνοεπιθέσεις, είτε είναι η τρομοκρατία τα οποία θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον, γιατί σε μεγάλο βαθμό ε, μας απασχόλησε το θέμα της ανταπόκρισης στην τρομοκρατία των τη τσιχαντιστική, εξτρεμιστική τρομοκρατία, χωρίς όμως αυτή να είναι η μοναδική απειλή. Και μην ξεχνάμε και την υποκίνηση του μίσους Πρόσφατα είχαμε ε, εκδηλώσεις από πλευράς της άκρας δεξιάς. Ε, επομένως θα πρέπει να έχουμε ένα πνεύμα ανοιχτό προς ε, η αδίποτε απειλή από όπου και αν προέρχεται άκρα δεξιά, άκρα αριστερά, τσιχαντιστικό εξτρεμισμό. Όλους αυτούς που προσπαθούν δηλαδή να ανατρέψουν, να διαταράξουν τον τρόπο με, οποίο, με τον οποίο έχουμε οργανώσει τις ζωές μας και ζούμε γενικά στις κοινωνίες μας και πιστεύω ότι και εσείς αυτό θα ε, συμβάλλετε πολύ. Πιστεύω ότι όταν ε, μελετούμε τις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ενσωμάτωση στις κοινωνίες μας, ε, τα προβλήματα τα σχετικά με την ενσωμάτωση και όταν, επί παραδείγματι, η... μας απασχολούν τα θέματα της ρεζοπαστικοποίησης ή της τρομοκρατίας, Οπωσδήποτε εσείς έχετε πολύ καλέ ιδέε για το πώς ε, μπορούν αυτά να αντιμετωπιστούν, τα εκφράζετε μέσω τη Επιτροπής σας και των εκθέσεών σας. Η Επιτροπή πάντως από πλευρά τη Επιτροπής πρέπει να σας πω ότι προσπαθούμε όποτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά να αποφύγουμε τον στιγματισμό ε, μιας συγκεκριμένης ομάδας ή τμήματος της κοινωνίας. Γιατί αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να ε, χρησιμοποιήσει βία ει βάρο των κοινωνιών μα είναι απλώς ένας κακός άνθρωπος, άτομο. Δεν, είναι, δεν εκπροσωπεί ούτε την κοινότητά του, ούτε τη θρησκεία του, εάν πρόκειται για θρησκευτικό εξτρεμισμό. Και πολύ συχνά ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτά τα κακόπιστα άτομα είναι η συνεργασία με την ευρύτερη κοινότητα. Και έτσι και προλαβαίνουμε εκείνον που ενδεχομένω να πέσει ένα πειρασμό να ακολουθεί τον δρόμο αυτό. Καταρχάς. Και δεύτερον, μπορούμε συνεργαζόμενοι με την κοινότητα αυτήν να ε, αντιμετωπίσουμε τα άτομα αυτά. Ανάλογα με τη χώρα έχουν δοθεί και διαφορετικές λύσεις. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τρόπου με τον οποίο ε, λειτουργεί η προσπάθεια για την καταπολέμηση τρομοκρατία και δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό, ότι μπορούν να μας βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό μην το λησμονείτε παρακαλώ, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που ε, πρέπει να έχετε υπόψη και για την εκθέσή σας. Επίσης, για το πώς μπορεί το Κοινοβούλιο να οργανωθεί στο μέλλον. Με συγχωρείτε, αλλά θα επιφυλαχθώ πάντω δικαιώματό μου και θα τηρήσω το δικαίωμα στη σιωπή. Ε, είναι αρμόδιο το Κοινοβούλιο να αποφασίσει. Και για την Επιτροπή βεβαίω και η Επιτροπή πρέπει να οργανωθεί και να, εξασφαλίσει του απαραίτητου πόρου και να στηρίξει το Κοινοβούλιο στον τρόπο τον οποίο θα έχει επιλέξει το Κοινοβούλιο για να οργανώσει τι εργασίε του. Για τα θέματα τη έκδοση ή για όλη αυτή τη συζήτηση για το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν του τελευταίου διαστήματο ε, θεωρώ απόλυτα πεπισμένο ότι όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να υπηρετούν το στόχο για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί. Και αν δεν τον υπηρετούν, προ τη μία την άλλη κατεύθυνση, θετικά ή αρνητικά. Δηλαδή, είτε χρησιμοποιούνται για λάθο στόχο, είτε δεν εξυπηρετούν ε, τον στόχο αυτόν για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί, τότε θα πρέπει να αντιδρούμε διότι διακυβεύεται η αξιοπιστία των εργαλείων αυτών, των μέτρων αυτών και όπως είπα πρέπει να υπηρετούν το στόχο που έχουν, για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί και μόνο αυτόν. Ε, στο θέμα της ε, υλοποίηση, ένα πράγμα θα πω. Συζητήσαμε και νωρίτερα μάλιστα πριν έρθετε εσείς, ε, συζητήσαμε το θέμα της υλοποίησης από τα κράτη-μέλη και θα παρακολουθήσουμε αυτή τους την πορεία για να βεβαιωνόμαστε ότι κάνουν ό,τι οφείλουν. Το θέμα δεν είναι όμως ότι μένουν, έχουν μείνει σε ένα σιρτάρι γραφείου και έχουν, έχουν αγνοηθεί αυτές οι οδηγίες. Απλώς ότι είναι πολύ συχνά δύσκολη η εφαρμογή τους στην πράξη. Και εκεί εντοπίζω εγώ τη δυσκολία. Αυτό πρέπει να προωθηθεί, όπω υπόθηκε νωρίτερα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει δηλαδή απουσία πολιτική βούληση και είμαι πεπισμένο ότι δεν υπάρχει απουσία πολιτική βούληση για την εφαρμογή του. Αλλά σε ορισμένε περιπτώσει η ε, μετατροπή σε πράξη αυτής της πολιτικής ε, βούλησης ε, έχει τους περιορισμούς της που οφείλονται και σε πρακτικέ δυσκολίε για τη νέα νομοθεσία δεν ε, διστάζουμε να προτείνουμε νέες, ε, νέα νομοθετήματα. Άλλωστε και στην ε, ομιλία για την κατάσταση ένωση τον προηγούμενο μήνα αναγγέλθηκε, εξαγγέλθηκε κάτι τέτοιο. Αλλά η πρόκληση πάνω απ' όλα είναι η υλοποίηση σε αυτούς όρους των όσων έχουν ήδη νομοθετηθεί και η εφαρμογή των συμφωνιών. Αυτή είναι η πρόκληση για το επόμενο εξάμεινο, για τους επόμενους μήνες. Είναι μεγάλη πρόκληση. Οι συνομοθέτες πρέπει να νομοθετήσουν πάνω με βάση τις προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί και μαζί με τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλιστεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και μετά εσείς μπορείτε να προσδορίσετε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο και να ορίσετε τα θέματα τα οποία θα κληθεί να συζητήσει το προσεχές κοινοβούλιο, προσεχής ε, σύνθεση. Όμως σε αυτή τη δουλειά μη και τα όσα έχουν να γίνουν σε πρακτικούς όρους για τους επόμενους μήνες, μέχρι τα τέλη του Μαρτίου, αρχές Απριλίου που έχουμε το νομοθετικό το περιθώριο της νομοθετική ε, εργασίας, θα έλεγα ότι κάθε μήνας μετράει, πρέπει να εστιαστούμε στην υλοποίηση όχι για να αποφύγουμε τη δυσκολία που θα, ήταν το να, που θα σήμαινε το να καλυφθούν άλλα κενά, η ενίσχυση της συνεργασίας, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το συζητήσω αυτό και μου φαίνεται ε, πολύ ευπρόσδεκτη αυτή η σχετική σας έκθεση, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να προχωρήσει η υλοποίηση. Για τους πόρους, οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει για την αντιμετώπιση της ε, διαδικτυακής διαγραμμικής ε, απειλής και νομίζω μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο εν προκειμένου ότι χρειάζονται και από πλευρά σα ή από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση πόροι, αλλά και από πλευρά των κρατών μελών. Πρέπει να διαθέσουν του απαραίτητου πόρου, γιατί δεν το πράττουν όλα τα κράτη-μέλη. Αν λοιπόν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε αυτό το μοντέλο, για τη συγκεκριμένη περίπτωση διαχρονική επιλύση, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε και στι άλλε υποθέσει με ε, ρητή υποχρέωση των κρατών μελών να διαθέσουν του πόρου όπως συμφωνούμε άλλωστε στις προτάσεις, όπως διατυπώνεται η συμφωνία τους και στις προτάσεις. Ε, Επίση, για την προσεχή δημοσιονομική περίοδο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώ ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι για την ε, ασφάλεια κατόπιν συζητήσεως με εσά και με τα κράτη-μέλη. Πάντως, εμεί προτείνουμε το διπλασιασμό της χρηματοδότησης για την εσωτερική ασφάλεια, τον τριπλασιασμό της ασφάλειας, των μέτρων που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα. Ειδικά έχουμε δύο εκατομμύρια στον ε, προϋπολογισμό καινοτομία για τη διαγραμμική απειλή, αλλά και στην έρευνα για την ε, ενσωμάτωση του, της έννοιας της ασφάλειας σε κάθε άλλο ε, ε, τμήμα του προπολογισμού όπω στη χρηματοδότηση για τι περιφέρειες κτλ. Να ενισχυθεί η ασφάλεια. Πάντω χρειαζόμαστε την δική σα υποστήριξη αλλά και των κρατών μελών και νομίζω ότι αν έχουμε τη δική σα υποστήριξη μπορούμε να έχουμε καλά παραδείγματα για προβολή. Για τη βάση δεδομένων δεν ήσταν να το είπαμε. Ίσως θα μπορούσαμε να το συνεχίσουμε διμερώς. Πάντω, εγώ θέλω να βρω έναν τρόπο για να προωθήσω την διαλειτουργικότητα Λαμβάνοντα υπόψη τι ανησυχίε που εκφράστηκαν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα να τα διεκπαιρεώσουμε στην τρέχουσα θητεία. Σα ευχαριστώ αγαπητέ Επίτροπε. Ευχαριστώ θερμά και για την διεξοδική ανάλυση που μας έκανες, για τη σαφήνεια με την οποία μίλησες και για τις πολύ ποιοτικές απαντήσεις που έδωσες και την έντιμη και ειλικρινή προπτική που επίσης που χάραξες ε, για τους επόμενους μήνες, ε, αλλά και πιο μακροπρόθεσμα. Ναι. Και ευχαριστώ και για την προθυμία σου να έρθεις. Εκ μέρους των συναδέλφων θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά, αλλά να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους, γιατί η εβδομάδα της Ολομέλειας ε, είναι πλήρη συνήθως στο πρόγραμμα φορτωμένο και είναι δύσκολο να έχουμε σε συνεδρίαση τέτοια παρουσία. Πάντως μην ξεχνάτε την επόμενη μας συνεδρίαση που θα γίνει στις Βρυξέλλες 9 Οκτωβρίου 9 με 12.30. Σα δίνω ραντεβού οπωσδήποτε ε, γιατί θα έχουμε ακρόση με τις τελικές αρχές αλλά θα εξετάσουμε και τις τροπολογίες ε, και τις συμβαστικές τροπολογίες ε, πάνω στις 1520 τροπολογίες οπότε έχουμε Πλήρε πρόγραμμα και στι 9 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ τον Επίτροπο και τη Γραμματεία, τη Λετήσια και ε, όλο το επιτελείο μας που κάνουν να μοιάζουν εύκολα πράγματα που είναι πολύ δύσκολα.